Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα παρακαλώ να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα τη συνεδρίασή μας. Χθε σας εξήγησα γιατί ξεκινάμε αντί για 9 στις 8.30. Ε, όπως είπαμε στις 11.30 θα έχουμε την πανηγυρική εκδήλωση για τον εορτασμό της 60ης υπετίου της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ρώμης. Περνάμε στις ψηφοφορίες. πρώτη ψηφοφορία αφορά τη γνωμοδότηση Νίκολσον, πρωτοβουλία για την αποδοτική χρήση των πόρων, μείωση της πατάλης τροφίμων και βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για γνωμοδότηση του κυρίου Νίκολσον. Αρμόδια κατ' επιτροπή είναι Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έχουμε ούκολες τροπολογίες και συμβαστικές επίσης τροπολογίες. Θα ήθελα να παρακαλέσω το συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Νίκολσον. Αν θέλει το λόγο, είναι η ώρα κύριε Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που βλέπω πόσοι ευρωπουλευτές ε, έφτασαν εδώ τόσο νωρίς το πρωί, φρέσκι φρέσκι, Νομίζω ότι πρέπει να επενέσω τον ενθουσιασμό που υπάρχει στην Επιτροπή μας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό μου καταρχάς και να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Ε, όσον αφορά την ε, εξέβρεση συμβαστικών προτάσεων ε, και νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρόταση για τη Γεωργία. Κύριε Πρόεδρε, θα αρκεστώ σε αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ καλά που θυμηθήκατε και τους συνεργάτες μας και τους βοηθούς μας, γιατί πραγματικά μας βοηθούν πολύ. Πάμε στην ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε ε, βάλει τις κάρτες σας. Ξεκινάμε. Τροπολογία 1. Διανατάσσεως της χειρός. Τις συμβαστικές τροπολογίες ε, ηλεκτρονικά. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 1, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Α. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, όπως είπα, τις συμβαστικές τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ο κύριος Άγνιου ζήτησε το λόγο. Ο κύριος Μποβέ μου λέει ότι δεν ε, χρειάζεται να βάλω τη κάρτα μου. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε, αλλά ούτως ή άλλως δεν φαίνεται να λειτουργεί. Να δοκιμάσω δίπλα. Δεν μπορώ να βάλω την κάρτα μου στη συσκευή. Λόγω του Brexit, λέει ο πρόεδρος. Brexit appears to have appeared premature. Το Brexit ε, νομίζω έφτασε πολύ νωρί. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να κοιτάτε το χέρι μου. Εγώ καταψήφισα πάντω τη συγκεκριμένη τροπολογία. Α, τώρα λειτουργεί. Ε. Παρακαλώ να σημειώσουμε την ψήφο του κυρίου Άγνιου. Ούτως ή άλλως δεν αλλάζει το αποτέλεσμα μία ψήφος κατά, αλλά τη σημειώνουμε. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία Β. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την συμβαστική Β. Τέλος ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Συμβαστική τροπολογία C. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ωραία. Ε, συμβαστική τροπολογία σε Α. Άρχεται η ψηφοφορία για την CA, ε, συμβαστική τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 της κυρίας Κέρστιγκερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D α μικρό Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία, όχι μάλλον τροπολογία 16, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ε ή άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 19. Διανατάσσεως της χειρός. Ποιο είναι υπέρ τη 19, εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ, εγκρίνεται. 84, 84 ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 41. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 43. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 44. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία F, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρο... Η συμβαστική τροπολογία. Πάμε στην τροπολογία 53. Ποιος είναι υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία G. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται όπως και 70 με την ίδια διαφορά. Συμβαστική τροπολογία H. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία J. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 116. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 117. Υπέρ. Κα... Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 121. 13 αποχή. Συμβαστική τροπολογία και Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία L. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία M. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται συμβαστική όμικρον. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική π. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Q. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Τροπολογία 131, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 132, ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 132, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. Τροπολογία 133. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. κοινή τροπολογία για το νερό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία για το νερό. Περνάμε στην 144. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 147. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 150. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 151. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 167. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 22 ήταν ψηφή κατά. 172. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Και ψήφο Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως έχει τροποποιηθεί, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση και συγχαίρουμε τον εισηγητή, τον κύριο Νίκολσον. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο για Κάποιο σχόλιο, όχι. Ε, στην 9 ε, ε, με 11 Απριλίου θα ψηφιστεί η έκθεση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα πάει στην Ολομέλεια του Μαΐου. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία της έκθεσης Νόιχλ. Αρκετά επιμαχό θέμα. Μάλιστα, είχαμε και την συμβολή εμπειρογνωμών από την Ολλανδία, αλλά αρμόδια να μας ενημερώσει καλύτερα η συγγήτρια, η κυρία Νόιχλ. Παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Γραμματεία και φυσικά τους σκιώδεις εισηγητές. Ήτανε πολύ επικοδομητικές οι συναντήσεις, ε, δεν είχαμε προβλήματα από κοινού και πολύ ομαλά ε, κάναμε τις εργασίες. Θα ήθελα να σας πω ότι μετά τη συμβαστική τροπολογία L, έχουμε μία πρόταση βελτιωμένη και βλέπετε εκεί που αναφέρεται η τροπολογία του εισηγητή. Ε, στο 3.20 και 3.18 ε, έχουν ε, αλλάξει το συν και το πλήν. Κατά τα άλλα πάντως, σας ευχαριστώ πολύ και για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Νόεχολ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία Α. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 152. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 152. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 153. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός ελεγχός για την 153 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 154. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. Συμβαστική τροπολογία Β. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Σ. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική C. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 188. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε στην 199 της συγγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. Τροπολογία 234. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 234 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία G. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 245. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 246. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 248. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 249. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 254. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 254. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Τροπολογία 258. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 259. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 260. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται αλλά στο ελέγξουμε καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 261 υπέρ. Υπέρ της 261. Εγκρίνεται. 263. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 264 υπέρ. Το κυρίου Ντες. 264. Κατά. Απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία I. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 277. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 277. Άρχεται ψηφοφορία. ψηφοφορία. Zamykamy głosowanie. Odrzucona. Απορρίπτεται. Ποιο είναι υπέρ τη 279 του κυρίου Μπράνεν. Κατά. Εγκρίνεται η 279 και πάμε στη συμβαστική τροπολογία J. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Ε, πάμε στη 294. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 294. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Κ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 312 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία λάμδα. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική L. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τροπολογία 318. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, δεν έχει δύο τμήματα, ενία είναι. Απλώς είναι δύο τροπολογίες μαζί, 318 και 319. Είναι πανομοιότυπε. υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία μη. Πρώτα όμω. ή ε, όχι, δεν θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για τις προηγούμενες τροπολογίες. Πάμε στη συμβαστική μη, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. Τροπολογία 331. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία νη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 της κυρίας Χόιμπουχ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία όμικρον. Αλλά πρώτα θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 345 Χόιμπουχ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία όμικρον. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 357. Και πάλι της κυρίας Χόιμπουχ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία π. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται 364 της κυρίας Πετήρ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 365 της ιδέας υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 της κυρίας Νόιχουλ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κανονικά γίνεται δεκτή, αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 της συγγήτριας, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 17, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 19 της συγγήτριας, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 33, ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 33, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 της συγγετρίας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 7. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 55 πάλι της ηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Για Εγκρίνεται τροπολογία συμβαστική υπαριθμών 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Ποιος είναι υπέρ της εκατοστής τροπολογίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 107. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 108 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 111. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά καλό κακό θα ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 13, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 123 και 124 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, γιατί ναι, μάλλον έχει εγκριθεί, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία παριθμό 14. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 130 της κυρίας Νόιχλ. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος όμως για την 133 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον εγκρίνεται πάντως άρχεται ψηφοφορία για την 137 τέλος εγκρίνεται 138 υπέρ εγκρίνεται και 139 υπέρ εγκρίνεται με την ίδια διαφορά, με την ίδια πλειοψηφία. Οπότε ψηφίζουμε το ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί. Ε, και τώρα Ελεκτρονικά το ψήφισμα με τις τροπολογίες. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεν ξέρω αν η κυρία Συγγετρία, η κυρία Νόεχλη θα ήθελε να σχολιάσει κάτι. Παρακαλώ. Ήθελα απλά να σας ευχαριστήσω Τώρα θα περάσουμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ τους Κιώδης. Ήταν πολύ επικοδομητική συνεργασία. Ε, ναι, ε, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από τα κράτη-μέλη για την έκθεση σας, κυρία Νόεχλου. Ε, θα περάσει στη δεύτερη ολομέλεια του Απριλίου, αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί, δεν είναι σίγουρο. Περνάμε στο σημείο 8. Ε, κατεξιοδότηση κανονισμού Επιτροπής για την τροπολογία του κατεξιοδότηση κανονισμού 639 του 2014 σχετικά με τα μέτρα ελέγχου για την καλλιέργεια κάναβης και ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού, τις ενισχύσεις αγροτών νεαρής ηλικία, οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο νομικού προσώπου, του υπολογισμού του αναμονάδα ποσού στο πλαίσιο της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα τμήματα δικαιωμάτων ενίσχυσης και ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίηση που σχετίζονται με το καθεστώς ενιαίας τρεματικής ενίσχυσης και την προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση καθώς και για την τροποποίηση του παραρτήματος 10 του κανονισμού υπαριθμών 1307 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πολύ περίπλοκη διατύπωση, αλλά νομίζω ότι ξέρουμε περί την πρόκειται. Πρόκειται για την έγκριση της σύστασης των συντονιστών της Επιτροπής Γεωργίας να ζητηθεί παράταση της δίμηνης προθεσμίας διατύπωση αντιρρήσεων. Παράταση κατά δίμηνο. Θα ψηφίσουμε τώρα, όπως θα θυμάστε, στις 9 Μαρτίου ε, είχαμε την διαδικασία, την γραπτή διαδικασία μέσω της γραμματείας για την ανατροπή της απόφασης των συντονιστών της άκρη της 28 Φεβρουαρίου και κατόπιν έγινε η διατυπώθηκε υποστήριξη ολόκληρης επιτροπής ε, να μην ζητηθεί παράταση κατά δύο μήνες της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεως στην κατεξοδότηση πράξη. Τελικά συμφώνησαν ε, οι περισσότεροι συντονιστές για το αίτημα δίμηνης παράτασης και μετά από συζήτηση που έγινε στην τελευταία συνεδρία στο Στρασβούργο 13 Μαρτίου, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Επιτροπής το αίτημα αυτό για δίμηνη παράταση. Τώρα θα ψηφίσουμε τη σύσταση των συντονισμών της Επιτροπής Γεωργίας να ζητηθεί παράταση της ε, δίμηνης προθεσμίας ε, ε, διατύπωσης αντιρρήσεων για ένα δίμηνο ακόμη. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, μια και δεν βλέπω να υπάρχουν ερωτήσεις. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, για την παράταση κατά ένα δίμηνο της προθεσμίας. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι ψηφίσατε όλοι. Οπότε, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η σύσταση των συντονιστών. Οπότε το 9 καταπίπτει δεν έχει νόημα να ψηφίσουμε. Έχουμε πλέον τη δίμηνη παράταση. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 10. Τη γνωμοδότηση της κυρίας Κάστιγκερ. Αλλά ζήτησε το λόγο ο κύριος Νίκολσον. Παρακαλώ. Ναι κύριε Πρόεδρε, Ήθελα να θέσω το εξή που ακούσαμε στην τηλεόραση τις τελευταίες δύο μέρες ε, για σάπιο βοδινό που εξάγεται από την ε, Βραζιλία. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι. Αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε τη γραμματεία, ποιος, ε, την Κομισιόν, ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε την ευθύνη να ρωτήσουμε. Έχει έρθει βόιο κρέα από τη Βραζιλία και έχει μπει σε κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. σάπιο μπορούμε να το εντοπίσουμε, να μας πούν πόσο, πού και πότε. Δεν θέλω να δημιουργήσω αναστάτωση, αλλά πιστεύω ότι αποτελεί ευθύνη μας να κάνουμε το ερώτημα και η Κομισιόν να ψάξει να το βρει και να μας δώσει μια απάντηση, αν είναι δυνατόν σήμερα, αλλιώ ε, κάποια άλλη στιγμή ή έστω και γραπτός ε, το συντομότερο δυνατόν. Ε, δεν ξέρω, ίσως να δούμε και ποια είναι η κανονική διαδικασία. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός με τους κανόνες και τις διαδικασίες, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να το ε, ε, υπογραμμίσουμε και να το θέσουμε ως ζήτημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνε ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω το αίτημα του κυρίου Νίκολσον προτείνω το εξή. Το απόγευμα, υπό το σημείο 13, θα έχουμε την ευκαιρία γιατί θα έχουμε εκπροσώπου τη Επιτροπή που θα μα μιλήσουν για εμπορικέ διαπραγματεύσει. Και δεδομένου ότι ανέφερε το ζήτημα ο Τζέιμς Νίκολσον, θα μπορούσαμε να του θέσουμε το ζήτημα αυτό. Ναι, Δύο-τρει μέρε κυκλοφορούν κάποιε τέτοιε φήμε για εισαγωγή ελιωμένου κρέατο από τη Βραζιλία. Ε, είχα κάποιες συζητήσει και με τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδία Παραγωγών Τροφίμων και είχα σκεφτεί να στείλω και γραπτή ερώτηση προ την Επιτροπή. Αλλά προτίμησα να το χειριστεί η Γραμματεία. θα πρέπει να δούμε με ηλεκτρονικό το χειδρομείο, με ηλεκτρονική ελογραφία, αν μπορεί να έρθει το απόγευμα ο Γενικός Διευθυντής της Άγκρη και να συμπεριλάβει και αυτό το θέμα στην παρουσίαση. Η Γραμματεία, επαναλαμβάνω, θα κάνει το σχετικό διάβημα προς την, Επιτροπή, την Γενική Διεύθυνση Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά αιτήματα τέτοιου τύπου, μπορούμε άτυπα να τα διαβάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως ε, να λάβουμε μια απάντηση σήμερα το απόγευμα, να λάβουμε κάποια σύντομη εξήγηση. Αλλά μια ερώτηση, κύριε Νίκολσον, εσείς αναφερθήκατε σε σάπιο κρέας. Αυτό μήπω είναι θέμα τη γενική διεύθυνση υγεία ή τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Σήμερα το απόγευμα θα έρθει ο κύριος Κλάρκ από την Γενική Διεύθυνση Άγκρη που θα μιλήσει για τις διεθνείς εμπορικές ε, διαπραγματεύσεις. Πιθανότατα να μπορεί να πει κάτι για τις εισαγωγές από την Βραζιλία, όχι όμως όσον αφορά την πτυχή της υγείας. Μήπως θα πρέπει να ε, επικοινωνήσουμε και με τη Γενική Διεύθυνση Σάντε. Όντως, ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καλέσουμε για κάποιον από την Σάντε την Διεύθυνση υγεία. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει κάποιο από τη Γενική Διεύθυνση Απλά ρωτώ, έχει εισαχθεί κάτι τέτοιο από τη Βραζιλία τα τελευταία δύο χρόνια, για παράδειγμα, και σε τι ποσότητε. Ε, δεν περιμένω να μπορούν να βρουν όλε τι πληροφορίε μέχρι σήμερα το απόγευμα, αλλά να μα δώσουν κάποιε γενικέ πληροφορίε. Ε, εγώ απλά σα μεταφέρω αυτά που άκουσα στην τηλεόραση. Δεν ε, προσπαθώ να κατηγορήσω κανέναν προτού να λάβουμε τις πληροφορίες, ε, αλλά ας λάβουμε τις αναλυτικές πληροφορίες. Άλλωστε βρισκόμαστε στην αρχή της υπόθεσης αυτής. Ο κύριος Μποβέ. Euh, ναι, δεν σχετίζεται με το εμπόριο, σχετίζεται κάπως με το εμπόριο βέβαια, αλλά τίθεται ένα πρόβλημα ε, αφού το συζητήσαμε πρέπει να το συζητήσουμε και με την Κομισιόν ε, το θέμα ότι η Αμερικανική Διοίκηση στις Ενωμένες ε, Πολιτείες αποκάλυψε είναι το απόρριτο από την αλληλογραφία της Μονσάντο που ήδη το 89 γνώριζε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της γλυφοσάτης και των σχετικών προϊόντων και των εκδόχων της ε, και ότι αυτό δημιουργούσε ένα πρόβλημα υγείας. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει λοιπόν μια συζήτηση με την Επιτροπή, ίσως και με την Επιτροπή ε, Υγείας και Καταναλώσης, αλλά να ακούσουμε και την ΕΦΣΑ και τον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Είναι πιστεύω βασικότατο διότι είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί γιατί πρόκειται για ένα προϊόν που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τους γεωργούς Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Είναι συγκλονιστικό, συγκλονιστικές αυτές οι αποκαλύψεις. Εμά, εμένα προσωπικά δεν με εκπλήσουν, αλλά πράγματι σήμερα αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός πραγματικού γεωργικού και υγειονομικού σκανδάλου. Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στις εισαγωγές από τη Βραζιλία. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Νίκολσον στο αίτημά του προς την Κομισιό να μας δώσει πληροφορίες. Πράγματι είναι στρέπλωση του ανταγωνισμού εάν ε, γίνεται δήλωση των ποσοτήτων 15 ε, μέρες ε, πιο αργά. Ε, και σίγουρα θα πρέπει να προσέξουμε οι γεωργοί μας ε, στην ε, Ευρώπη να μην βρεθούν σε δυσχερέστερη θέση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ο κύριος Χόισλινγκ, ναι, όσον αφορά τη Βραζιλία, φυσικά θα πρέπει να σταματήσουμε τις εισαγωγές ε, τέτοιου κρέατος. Είναι θέμα όμως με σημαντικές επιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τις διαπραγματεύσεις Mercosur. Και ο Νίκολσον έχει απόλυτο δίκιο. Ισχύουν άλλα πρότυπα για τους ευρωπαϊκούς παραγωγούς. Θα πρέπει να φροντίσουμε και κατά τις εισαγωγές να τηρούνται τα ίδια πρότυπα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Σίγουρα πάντως θα πρέπει να θέσουμε ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Όντως, πολύ σημαντικό το θέμα και συμφωνούν ε, μεταξύ τους ακόμη και οι κύριοι Χόισλιν και Ντες. Να υπογραμμίσω αυτά που είπε ο κύριος Χόισλινγκ. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μιλήσουμε και με την DigiTrade για να δούμε τι θα κάνουμε με τις εισαγωγέ από τη Βραζιλία. Γιατί ε, ε δεδομένου ότι και εμεί δεν μπορούμε να εξάγουμε κρέα στη Βραζιλία. Ευχαριστώ κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως βλέπουμε μας καθησυχάζει η συζήτηση αυτή για κάποιες θέσεις που έχουμε λάβει ορισμένοι από εμά για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Περισσότερο από πουθενά αλλού πρέπει να προσέχουμε τον τομέα της γεωργίας. Να ζητήσουμε λοιπόν από την Κομισιόν διευκρινήσεις για αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με το ζήτημα της Βραζιλίας. Ε, άκουσα και τα όσα είπε ο κύριος Μποβέ, υποχρεούμεθα ουσιαστικά να κάνουμε μια συζήτηση με την ΕΦΣΑ για το ζήτημα των μελετών και των ελέγχων. Και η κυρία Αγγελέρα θα είναι η τελευταία σε αυτό το γύρο. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη η πρόταση του κυρίου Νίκολσον για σχετική συζήτηση. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στους ε, ελέγχους της εισαγωγές, σοβαρότατο πρόβλημα. Και έχουμε με το α ή το β προϊόν κατά καιρούς προβλήματα. Και μάλιστα είναι ανησυχητική η κρίση που επισήμαναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δεν έχουμε στοιχεία για τις ποσότητες που εισήχθησαν στην Ευρώπη, για το τι έχουμε καταναλώσει ή θα καταναλώσουμε και την τρώμε από τη Βραζιλία. Θα πρέπει νομίζω περισσότερο στην, ε, από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας ε, να ζητήσουμε εξηγήσει και όχι από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για να ενισχυθούν οι έλεγχοι στι αγωγέ. Είναι θέμα δημόσιας υγείας αυτό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είδος, τι τμήμα των παραγωγών αυτών έχουμε ήδη καταναλώσει, έχουμε ήδη φάει ή θα φάμε. Και είναι πολύ σημαντική η ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Άντε, εδώ, της ε, Διεύθυνσης Υγείας. Νομίζω ότι Υπάρχει ομοφωνία. Όλες ε, οι πολιτικές ομάδες ε, και σύσσωμη η Επιτροπή Γεωργίας ε, ζητούν εξηγήσει από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας. Θα στείλουμε τις σχετικές προσκλήσεις και στις δύο Γενικές Διευθύνσεις, Γεωργίας και Υγείας, από τη Γραμματεία και δεν ξέρω πότε θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Να σας πω κάτι, συντομία που μπορεί να ενδιαφέρει σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν στις 11 Απριλίου έχουμε οργανώσει συζήτηση σε αυτή την Επιτροπή με εκπρόσωπο της ΕΦΣΑ για οποιοδήποτε θέμα μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε στα γεωργικά θέματα και που αφορούν τις δραστηριότητες της ΕΦΣΑ στις 11 Απριλίου. Καλώς. αλλά και το σημερινό θέμα που επισήμανε συνάδελφοι είναι σημαντικό και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ε, εξηγήσει ε, που θα ζητήσουμε από τις Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας και Υγείας. Ωραία, περνάμε όπως είπα στο σημείο 10 τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, ε, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομεία ε, στο πλαίσιο ε, για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και τροποποίηση του κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου υπαριθμών 525 του 2013 με θέμα το μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Ε, η συγγήτρια εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας είναι η κυρία Κέρστιγκερ που συνέταξε την γνωμοδότηση. Αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι επιτροπή περιβάλλοντος. Εισηγητής είναι εκεί ο κύριος Νόρμπερτ Λίνς. Όπως είπα είναι αρμόδια επί της ουσίας αλλά ευτυχώς πολλά μέλη της Επιτροπής Γεωργίας είναι και μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, οπότε θα ακουστεί και εκεί έντονα η φωνή μας.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 ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των δασών και ε, γι' αυτό είναι σημαντικό που συζητάμε την ε, έκθεση αυτή σήμερα. Πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ε, όσον αφορά το πακέτο για το κλίμα και τις εκπομπές που έχουμε μπροστά μας. Καταρχάς, μια γενική παρατήρηση η επισητιστική ασφάλεια και η ε, βιώσιμη χρήση των πρώτων υλών δεν ε, αντίκειται στην πολιτική για το κλίμα. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ε, κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού. Επίσης, για μένα είναι σημαντικό να έχουμε συνεκτική προσέγγιση και να έχουμε και τόλμη για αλλαγές. Η γεωργία και η δασοκομεία ε, έχουν, ε, παίζουν εδώ ιδιαίτερο ρόλο, διότι αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε την ε, σύνδεση ανάμεσα στους τομείς αυτούς και να εκμεταλλευτούμε τις συνέργειες, αυτό θα είναι πολύ κρίμα. Και η προστασία του κλίματος είναι ένας τομέας ιδιαίτερης σημασίας. Για μένα είναι σημαντικό να πούμε ότι η γεωργία και η δασοκομεία αποτελούν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για τη Λουλουσιεφ και για μένα ήταν σημαντικό να επικεντρωθώ σε τρεις αρχές. Καταρχάς δικαιοσύνη, δεύτερον συγκρισιμότητα και ε, υποκατάσταση. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, είναι σημαντικό ε, τα αποτελέσματα που έχουν ήδη πετύχει τα κράτη-μέλη να μην ε, χρησιμοποιηθούν εις βάρος τους. Ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν επιφέρει τεράστιες βελτιώσεις στον τομέα της δασοπονίας. Και έχουμε κάποια κράτη-μέλη που εδώ και δεκαετίες εφαρμόζουν μέτρα για το περιβάλλον και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Η δεύτερη αρχή είναι η αρχή της συγκρισιμότητας. Εδώ με ενδιαφέρει κυρίως η αναδάσωση και η βιώσιμη δασοκομεία να ε, εκτιμηθούν θετικά. Υπάρχουν ε, σημαντικές διαφορές στα δάση της Ευρώπης από τη Φιλανδία μέχρι την Ελλάδα και δεν επιτρέπεται να τρέφουμε την αυταπάτη ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. One size fits all. Η τρίτη αρχή είναι η αρχή της αντικατάστασης και θα πρέπει εδώ να κάνουμε σαφή διάκριση ανάμεσα σε πράσινες, σε πράσινα καύσιμα και ορυκτά καύσιμα. Εάν δεν καταφέρουμε να κάνουμε την διάκριση, Ε, και να συνυπολογίσουμε και την ε, χρήση της ξυλίας, ε, για παράδειγμα, στις οικοδομές και αλλού. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίσουμε, διότι αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές. Και έχω ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα που είναι το τριπλό αποτέλεσμα ενός σπιτιού από ε, ξύλο, ότι αφενός αποθηκεύεται διοξίδιο το άνθρακα εκεί, αντικαθιστά ε, άλλα υλικά όπως είναι το τσιμέντο που χρειάζονται πολύ ενέργεια και τέλος μπορεί να ανακυκλωθεί το σπίτι και ασχολούμαστε τώρα με το πακέτο της ε, κυκλικής οικονομίας ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας. Αυτό λοιπόν είναι στην πράξη κυκλική οικονομία και για μένα είναι σημαντικό. Εδώ να καταλάβουμε όλη την αρχή αυτή. Συνοπτικά, όσον αφορά τη γνωμοδότησή μου, αυτό σημαίνει ότι θα πετύχουμε θετικά αποτελέσματα Εάν μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τον τομέα LULUCF στο πλαίσιο της κλιματικής πολιτικής, ε, πρέπει να εφαρμόσουμε μια πολιτική από τη βάση προς τα πάνω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επιτρέπεται να αλλάξει μόνη της ε, το επίπεδο αναφοράς των δασικών εκτάσεων. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, συμπεριλάβουμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα της βιοοικονομίας, να αναγνωρίσουμε δηλαδή τον τομέα αυτών και την ε, ανισορροπία ανάμεσα στη δεσοκομεία και την αναδάσωση να την ε, αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, θα πρέπει ε, να αναδοσώνονται οι περιοχές που, που αποψηλώνονται. Επίσης, θέλουμε βιώσιμη διαχείριση και δεν θα πρέπει να τιμωρείται αυτή, αντιθέτως θα πρέπει να αναγνωρίζεται. Θα είναι παράλογη η πολιτική μας εάν δεν καταφέρουμε να ανταμείψουμε τους τομείς που ήδη έχουν καταφέρει θετικά αποτελέσματα. Εάν, θέλουμε να δώσουμε, εάν καταφέρουμε να δώσουμε ένα σημαντικό κίνητρο για την πράσινη οικονομία και να μπορέσουμε σιγά σιγά βαθμιαία να μειώσουμε τις ορυκτές πηγές ενέργειας, τότε σίγουρα θα έχουμε κάνει κάτι σωστό. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία με τους ε, συναδέρφους εδώ στην Επιτροπή, αλλά και με την ε, εισηγήτρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα όραμα μακριά από τις ορυκτές πηγές ενέργειας ε, στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό και ότι στον τομέα LULUCF ε, μπορούμε να θέσουμε τις πρώτες κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να ακούσω ε, τα όσα έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Όπως θα θυμάστε, η κυρία Κώστιγκερ ετοίμασε και τη στρατηγική για τα δάση τη σχετική έκθεση, δηλαδή κάτι που φάνηκε και από τη γνωμοδότησή της. Χρειάστηκε να κάνει επιπλέον μαθήματα, έμεινε σαν να έμεινε μεταξυταστέα στα δάση και έπρεπε να επαναλάβει τη γνωμοδότηση για το Λουλουσιεφ. Πάντως είναι περίπου το θέμα και τα χρήσιμες γνώσεις από την προηγούμενη στρατηγική για τα δάση. Περνάμε τώρα στη συζήτηση. Ποιος θέλει το λόγο? Η κυρία Μίλλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ελίσαπετ Κρέστινγκερ για τη θέση που λαμβάνει όσον αφορά τα δάση, τους δασοπόνους και το πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ε, την πολλαπλή λειτουργικότητα των δασών ε, στην Ευρώπη. Προστατεύεται η βιοπικιλότητα, ε, βελτιώνεται το, η ποιότητα ζωής και ξέρουμε ότι εκμεταλλευόμαστε ε, το 65% μόνο των δασών, δηλαδή 35% των δασών αυξάνονται χωρίς να τα εκμεταλλευόμαστε. Παίζουν ε, λοιπόν ε, πολύ σημαντικό ρόλο ε, στην δέσμη αυτήν μέτρων τα δάση. Πρέπει να ενισχύσουμε τα δάση, την δασοπονία, διότι αυτό μακροπρόθεσμα είναι η καλύτερη στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας σε συμφωνούμε πάνω στο θέμα αυτό. Όσον αφορά το ΛΟΛΟΣΙΕΦ έχουμε τεράστια προβλήματα όσον αφορά τον υπολογισμό των επιπέδων αναφοράς των δασών των δασικών εκτάσεων. Δεν ε, υπάρχει εδώ πρόσθετη γραφειοκρατία για τους ε, δασοπόνους. Ε, φοβάμαι όμως ότι... τελικά θα έχουν σημαντικότερο άκτος οι δασοπόνοι από ό,τι μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα πρέπει εδώ από την πίσω πόρτα να ε, πετύχουμε παρέμβαση του ευρωπαϊκού επίπεδου, θα πρέπει να διατηρήσουμε την αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει να έχουμε μέτρα λοιπόν για την ε, προστασία του περιβάλλοντος ε, από πλευράς των δασοπόνων και θα πρέπει να είναι εφικτά και πρακτικά τα μέτρα αυτά. Έχουμε εδώ τρεις διαφορετικές θέσεις. δεν θα, έχουμε αφενός τη γεωργία, την δασοκομεία. Ε, δεν θα ήθελα όμως ε, να αποκλείσουμε εδώ και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Κυρία την στο πλαίσιο ε, των διαβουλεύσεων δεν ζητήσατε ομάδα εμπειρογνωμόνων. Ε, θα το προτιμούσα αυτό όμως από ε, την πρόταση του κυρίου Λίνς. Θα υποβάλουμε τροπολογίες και σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, θετική γνωμοδότηση για τα δάση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Με ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Και εγώ είμαι σκιώδης στην Επιτροπή ΕΝΒΗ Προσπαθώντας να καταλάβω το όλο θέμα, να καταλάβουμε το όλο θέμα, κάναμε μια διάσκεψη, μιλήσαμε με αγρότες, ε, ε, συνεργάστηκα με έναν περιβαλλοντολόγο μέλος του Πράσινου Κομματός ε, στο δικό μου κόμμα και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο υπολογισμός είναι ουσιώδου σημασία για να κάνουμε κάτι για τα αερία θερμοκήπη και την βλάβη προς το περιβάλλον και το κλίμα. Τα προβλήματα που διαπιστώσαμε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι αγρότες ε, και κάτι που μας ανησυχεί είναι ότι η δασοκομεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ιρλανδία για να αντισταθμίσει την πιο εντατική γεωργία και θα έλεγε κανείς ποιο είναι το πρόβλημα με όλα αυτά ουσιαστικά αυτό που ανησυχεί πολλού αγρότε με του οποίου συζητήσαμε είναι ότι υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί μια κατάσταση όπου η χειρότερη ε, γη, όπω την ονομάζουν ορισμένοι, η ορεινή γη, η αλληγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φυτευτούν δάση. Και έτσι οι περιοχές στο νότια της χώρας που είναι οι καλύτερες γεές θα προχωρήσουν με την εντατικοποίηση. Σε αυτό μπορεί να αρέσει, αλλά θα δημιουργήσει πρόβλημα στις περιοχές όπου ζω εγώ. Διότι θα έχει ως αποτέλεσμα βρία δασοκομεία σε πολλά εκτάρια και η εμπειρία μας λέει ότι αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να τους προφυλάξουμε λοιπόν. Και τι άλλο πρέπει να προφυλάξουμε. Ε, πρέπει να προφυλάξουμε το λαό μας από την ιδέα ότι ε, θα φυτευτούν δάση σε κάποια κακή γη. Και αντί να δεσμεύουμε άνθρακα ε, στην δασοπονία τα δέντρα δεν θα μεγαλώσουν καλά όπως θα βλέπουμε ε, λόγω των ανέμων και θα καταστρέψουμε ουσιαστικά τις καταβόθρες άνθρακα. Ε, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό. Θα έχει και αποτελέσματα για τους λαούς μας. Κάτι άλλο, συμφωνώ με το να χρησιμοποιούμε τους βάλτους, τους υγρότοπους. Το να γίνει αυτό υποχρεωτικό, από την εμπειρία μου ξέρω ότι δεν είναι καλή ιδέα. Το, θα το υποστήριζα αλλά ξέρω ότι δεν είναι καλό. Αν πάμε και πούμε στον κόσμο ότι οι γέες αυτές είναι πολύτιμες ε, ως καταβόθρες άνθρακα, όπως ε, λένε στου ανθρώπου στο Δουβλίνο ότι οι γέες πάνω στις οποίες ζουν ε, που κοστίζουν ένα σωρό λεφτά το στρέμα πάρα πο... είναι πολύτιμες οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν σε αυτές τις περιοχές ε, τις ε, θεωρούν ότι οι περιοχές αυτές είναι πολύτιμες και η ιστορία και το παρελθόν μας λέει ότι η αξία αυτή δεν κληρονομείται ε, και τελικά διότι ο κόσμος φεύγει από τις περιοχές αυτές γιατί είναι πιο δύσκολη διαβίωση εκεί. Χθες μόλις είδαμε ένα παράδειγμα κακής διαχείρισης και μην με παρανοήσετε, είμαι υπέρ αλλά πρέπει να έχουμε και τους ανθρώπους να μας υποστηρίξουν με την οδηγία για του οικοτόπου αλλά και για την πρόληψη τη κλιματική αλλαγή. είχαμε χθε στην Ιρλανδία μια κατάσταση όπου μια μικρή επιχείρηση ε, την έσυρα στα δικαστήρια και υπάρχει περίπτωση να λάβει πρόστιμο μισού εκατομμυρίου ε, ευρώ και να ε, τριετή φυλάκιση ε, και νομίζοντας έτσι ότι θα τους σταματήσουν να κάνουν αυτό που κάνουν αλλά ουσιαστικά θα κάνει όλους σε αυτό που κάνουμε εδώ. Θα μαυρώσει το όνομα των υποστηρικτών του περιβάλλοντος. Οπότε για να κάνουμε κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε μαζί μας και τους ψηφοφόρους μας και τους υπόλοιπους. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να λέμε ε, περάστε, σε κάποιον, περάστε τρία χρόνια στη φυλακή αν δεν κάνετε αυτό που λέμε. Πρέπει να τους πείσουμε. Και ουσιαστικά αυτό κάνω εγώ και άλλοι άνθρωποι στη χώρα μου αυτό προσπαθούν να κάνουν ώστε οι που προσπαθούμε να προφυλάξουμε να προφυλαχθούν διότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί θα τις προφυλάξουν και όχι επειδή εμείς ε, φυλακίζουμε κάποιον για τρία χρόνια ε, και το επιβάλλουμε ένα πρόστιμο ε, μισού εκατομμυρίου ευρώ και έχουμε ξαφνικά έναν, άγρο, έναν θυμωμένο αγρότη τρομα, κρατημένο για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Αυτό δεν θα τους αποτρέψει κάθε φορά που θα βλέπουν άνθρωπο που υποστηρίζει το περιβάλλον θα στρέφονται εναντίον του. Οπότε πρέπει να έχουμε με το μέρος μας αυτούς τους ανθρώπους και έτσι πρέπει να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος και να σταματήσουμε να κάνουμε αυτά που γίνονται στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Θα σας παρακαλούσα πάντως να μην μιλάτε περισσότερο από ό,τι μίλησε η ίδια συγγήτρια στις παρεμβάσεις σας, αν γίνεται. Και να καλωσορίσω και τους επισκέπτες α, ε, της κυρίας Μίλλερ. Σας καλωσορίζω θερμά. Τους καλεσμένους κυρίας Μίλλερ. Ο κύριος Αντριέ. πρώτο ο κύριος Αντριέ και μετά ο κύριος ε, Άγνιο, δεχομένως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Κέστιγκερ για την παρουσίαση της γνωμοδότησης. Ε, συμφωνώ μαζί της, γιατί το θέμα είναι όντως τεχνικό, φάνηκε και από την παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Συμφωνία των Παρισίων και λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο δυναμικό που έχει μετριασμού ο γεωργικός τομέας, το λέει η γνωμοδότηση. Και συμ... θεωρώ ότι και η Γεωργία θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Και γι' αυτό θα πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να συνυπολογίζουμε τις εκπομπές και την απορρόφηση από τη χρήση των γεών ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη γεωργία και τη δασοκομεία. Επίσης, ε, ε υπάρχουν πολλές αδυναμίες ε, στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά, την συνεισφορά του δασοκομικού κλάδου που συμβάλλει τα μάλα στην αηφορία της οικονομίας. Και έτσι όχι μόνο θα περιορίσουμε τον κίνδυνο να έχουμε αρνητικά υπόλοιπα στον κλάδο για τη χρήση της γης, αλλά θα επιτρέψουμε και μεταφορές κονδυλίων σε ό,τι αφορά το, την πτυχή ε, του κεφαλαίου 8 για τα δάση, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα επίπεδο αναφοράς που θα λαμβάνει υπόψη κάποια σχέδια αναβάθμισης και αηφόρου διαχείριση των δασών που γίνονται από τα κράτη-μέλη. Επίσης, χρήσιμο είναι να διευκρινίσουμε το ρόλο των επιμέρους κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση ενός επίπεδου αναφοράς για τα δάση. Κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να ε, επιφορτιστεί με, την, ε, με τον προσδιορισμό του επίπεδου αναφοράς, γιατί έχει την τεχνική και πολιτική ευθύνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη της εξασφάλισης της διαφάνειας της όλης διαδικασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Άγνιο. Πρέπει να επενθυμίσουμε στην Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα στην δασοκομεία, στα κράτη-μέλη. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Ο κύριο Φλάνναγκαν δεν πρέπει καν να ανησυχεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θέλει να φυτέψει δέντρα στην Ιρλανδία. Δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκλεγμένη κυβέρνηση τη Ιρλανδία, αν θέλει να ε, φυτέψει δέντρα επειδή κάποιο σέπισε, ε, είναι δικό του θέμα. Εγώ θέλω να μιλήσω για, το, για τα ξύλινα σπίτια. Πολλοί αγρότες στη Βρετανία απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ξύλινους φράχτες. Λένε ότι είναι κακό για το περιβάλλον και έτσι οι φράχτες ε, ε, τους έβαζαν πάνω ένα ελαφρύ χημικό και τώρα όλοι αυτοί οι φράχτες ε, σαπίζουν και το βλέπουμε στην περιοχή μου. Πέφτουν παντού αν είναι να, να χτίζει κανείς ξύλινα ε, σπίτια και βάζει τέτοιες ε, πασάλους στο έδαφος, πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Αλλιώς τα ε, σπίτια θα γκρεμίζονται μετά από μια δεκαετία, διότι υπάρχουν τα έντομα από το έδαφος που τρώνε, κατατρώνε το ξύλο αυτό. Τώρα αυτό που βλέπω εγώ στο σημείο 10, την πέμπτη γραμμή, παρακολουθήσει και έκθεση ε, για τα συστήματα ε, εκπομπών. Ας δούμε το δικό μου αγρόκτημα. Εγώ πρέπει δηλαδή να εκτιμήσω πόσο διοξίδιο του άνθρακα εκπέμπουμε, δηλαδή από όλα τα τρακτέρ που χρησιμοποιούμε και όλα τα άλλα διζελοκίνητα οχήματα που έχω στο αγρόκτημα. Μετά πρέπει να βρούμε τη φωτοσυνθετική ε, ποσοστή όλων των ε, φυτών εκεί. Πρέπει να έχουμε ένα νούμερο και γι' αυτό. Είναι ημερήσιο, εβδομαδιαίο, ετήσιο, ένα θεός ξέρει. Μετά πρέπει να δούμε πόσο μεθάνιο εκπέμπουν τα πρόβατά μας. Και αυτό ποικίλει, είναι μεγάλα, είναι αρνιά, τι τρώνε. Ε, τρώνε ε, συσσωματώματα, πρέπει, κάποιος δηλαδή, πρέπει να τα αποφασίσει όλα αυτά και να τα γράψει κάπου και μετά πάμε στο οξύδιο του αζότου από τα ψυχανθή. Και αυτό πρέπει να το υπολογίσουμε. Αυτά που μεγαλώνουν κανονικά εκπέμπουν περισσότερο άζωτο και άλλα που δεν ε, ε, που είναι γεμάτα μήκητες ε, και ζυζάνια εκπέμπουν λιγότερο. Αυτό ζητάτε από τους αγρότες. Δεν βλέπετε ότι είναι αδύνατον να αρχίσει κανείς να τσεκάρει τετραγωνάκια ε, ε, για όλες αυτές τις πληροφορίες δεν πρόκειται να μας οδηγήσει πουθενά αυτό. Ευχαριστώ. Καπούτο. Κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη συναδέλφο κυρία Κώστιγκερ για την εξαιρετική της δουλειά και τις τροπολογίες που συμμερίζομαι. Η ενσωμάτωση του LULUCF στην πολιτική προστασία του κλίματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 πιστεύω είναι σημαντική συνιστόσα για μια σωστή ευστοχή ε, κλιματική πολιτική ε, και υπέρ τη βιωσιμότητα. Ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία. Θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι είναι αναγκαίο όχι μόνο να βασιστούμε στις, στα θετικά αποτελέσματα της προστασίας του κλίματος μέσω ε, μέτρων αναδάσωσης, αλλά να γνωρίζουμε και τι δυνατότητε του μετριασμού των κλιματικών επιπτώσεων μέσω της διαχείριση των δασών και της χρήσης ε, ε, βιώσιμων βιομαζών. Θεωρώ δεύτερον ότι η χρήση των βιομαζών ε, που είναι βιώσιμες και η ασφάλεια ενεργειακής ε, τροφοδοσίας, αναγκαιακού αφοδιασμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα κριτήρια για τις τιμές αναφορές, ε, αναφοράς για τα δάση στα κράτη-μέλη και τρίτον Όπως έχω ήδη πει στην έκθεσή μου για τον ε, επιμερισμό προσπαθειών, πιστεύω ότι η κατεξουδότηση πράξης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τροποποίηση των ε, κομματιών της βασικής νομικής πράξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει κυρία Πετήρ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κέστιγκερ για την πολύ αξιόλογη γνωμοδότησή της και να συμφωνήσω με την προσέγγισή της. Βέβαια, σε ό,τι αφορά το Λουλουσιεφ, ε, δύο ανησυχίες έχω και θα ήθελα να με στηρίξει και η συγκεκριμένη στο σημείο 8 Αναφέρεται ο τρόπος ε, υπολογισμού των ε, ε, καυσαερίων και αναφέρεται ότι το νέο επίπεδο αναφοράς θα προσδιορίζεται με βάση τις μέχρι τώρα πρακτικές, την ένταση διαχείρισης των δασών και με στοιχεία από το 1990 ε, βέβαια, από το 1990 μέχρι ε, το 1998, σε, για μεγάλο τμήμα, τα κρατικά δάση ήταν υπό την κατοχή των, ε, του Ιουγκοσλαβικού στρατού, οπότε είχε ε, αλλάξει η διαχείριση σε σχέση με το 2001-2013 ήταν πολύ διαφορετική η ένταση διαχείρισης ε, σε ό,τι αφορά τη δεκαετία του 90 και, το 2000, ε, και τη δεκαετία του 2000. Οπότε η περίοδος αναφοράς που προτείνεται είναι απαράδεκτη για την Κροατία, γιατί τότε δεν είχαμε δυνατότητα πρόσβαση στα δάση, γιατί ήταν υποκατοχή γιουγκοσλαβική. Και μάλιστα λαφυραγωγήθηκαν οι περιοχές αυτές χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση από τη Σερβία στην Κροατία. Ήταν επίσης ε, πολύ σημαντικές οι αρνητικές συνέπειες ε, του πολέμου για την Κροατία. Υποβαθμίστηκαν ε, οι δομές ε, στα δάση, είχαμε αποψήλωση των δασών, είχαμε απερίμωση των περιοχών, οπότε θα ήθελα να ληφθεί υπόψη αυτή η ιδιαιτερότητα και να ληφθεί υπόψη το αίτημα της Κροατίας. Ελπίζω να με υποστηρίξει η Επιτροπή Γεωργίας και η Συγήτρια. Επίσης, αυτή η πρόταση κατά τη γνώμη μου είναι άδικη γιατί ε, ουσιαστικά τιμωρούνται τα κράτη που κάνουν αηφόρο διαχείριση των δασών τους. Γιατί χώρες που είχαν πολύ αηφόρο διαχείριση δεν ε, εποφελούνται από την ελαστικότητα που προτείνει το Λουλουσιεφ. Μάλιστα, η Κροατία έχει 25% εκπομπές στο τομέα εκτό ε, του ETS και αυτή την ε, ευελιξία μπορεί να την αξιοποιήσει μόνο στο 0,5%. Και μάλιστα, δεδομένη τη μεγάλη έκταση των δασών στην Κροατία, εμεί δεν έχουμε στην Κροατία μεγάλη δυνατότητα περαιτέρω αναδάσωση. Οπότε και μάλιστα όλες αυτές οι μέχρι τώρα ε, περιοχές ε, στην ε, Κροατία ούτως ή άλλως εντάσσονται στο Natura 2000 στο οικολογικό δίκτυο που δεν επιτρέπει αλλαγή χρήσης γης. Οπότε έχουμε και πάλι διακλαδικό διατομιακό πρόβλημα στην Κροατία. Γιατί η συνολική επιφάνεια της Κροατίας που εμπίπτει στην Natura 2000 δεν μπορεί να αλλάξει σε ό,τι αφορά τη χρήση γης. Και επίσης αυτό είναι, αναφέρεται σε ένα ποσοστό 36%. Επίσης είχαμε ε, μείωση ε, το 2012, 38% ε, ε, μείωση των εκπομπών και συνολική, συνολική μείωση εκπομπών 21%. Και μάλιστα η μείωση των εκπομπών στην Κροατία οφείλεται στην μείωση του ζωικού κεφαλαίου των αγελάδων. Κάτι που έχει πολύ αρνητικέ συνέπειες στις γεωργικές εκτάσεις. Οπότε έχουμε πρόβλημα με την πρόταση αυτή. Και μάλιστα στις χώρες μέλη που διασφαλίστηκε μία βιοπικιλότητα Δυστυχώς ε, δεν επιβραβεύονται οι χώρες αυτές από τη συγκεκριμένη πρόταση και θεωρώ ότι αυτή η ιδιαιτερότητα των κρατών μελών ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την γνωμοδότηση και από την σχετική έκθεση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Χόισλινγκ. Ναι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Κρέστινγκερ για την έκθεση. Θα ήθελα όμως να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις ε, προς μια άλλη κατεύθυνση. Ε, υπόθηκε ότι δεν θα πρέπει να εξοραίζουμε την κατάσταση. Ε, πολύ μικρό μέρος ε, του θέματος είναι η προβληματική για το κλίμα. Η παραγωγή ενέργειας ε, από όλα τα δάση της Γερμανίας ε, αντιστοιχεί ε, στο μεγαλύτερο ανθρακοριχείο της Γερμανίας και θα πρέπει διασυνοριακά να σκεφτούμε διότι Μπορεί κάποιο να θεωρήσει ότι αφού έχουμε δάσο σε μία χώρα, στην άλλη χώρα μπορούμε να ε, ρηπαίνουμε όσο θέλουμε. Θα πρέπει να εξετάσουμε συνολικά το θέμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Επίσης, όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Κέστιγκερ. Η χρήση ξυλίας επί της αρχής είναι ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά είναι και κάπως αφελές να πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει καθόλου να υπολογίζουμε τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Τελείως ουδέτερη δεν είναι ούτε η βιοενέργεια. Επίσης υπόθηκε ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς, έχουμε άλλες καταβόθρες εξιδίου του άνθρακα όπως είναι η βάλτη. Θα πρέπει φυσικά να το σκεφτούμε και αυτό. Η βάλτη ε, είναι η μεγαλύτερε ε, καταβόθρες οξυδιού του άνθρακα στην Ευρώπη. Και όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριο Άκνιου, ότι ε, τα ξύλινα σπίτια τα τρώνε τα έντομα, η οικογένεια μου έχει ξύλινο σπίτι από το 1650. Πάντα εκεί κατοικούσαμε, χωρίς χημικά. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί το ξύλο επί πάνω, επί 100 χρόνια. Δεν ξέρω τι γίνεται στη δική σας χώρα, στη Γερμανία πάντως ε, είναι δυνατόν. Και φυσικά ε, είναι σκόπιμο να χτίζουμε ξύλινα σπίτια διότι δεσμεύεται έτσι το διοξείδιο του άνθρακα και αντικαθίσταται το βετό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά την Ελίσα Πετκόστινγκερ για την πρόταση που μας υπέβαλε, την οποία μπορεί να στηρίξει η πολιτική μου ομάδα. Χαίρομαι πολύ που η κυρία Κέρστιγκερ έχει αναλάβει την έκθεση αυτή. Όπως όλοι γνωρίζουμε, προέρχεται από την Αυστρία και έχει πολύ βιώσιμη δασοκομεία η Αυστρία. Ε, αγαπητέ Μάρτιν Χόισλινγκ, ε, όταν ε, δεν ε, λέμε άσχημα πράγματα, όταν δεν κατηγορούμε την κατάσταση, δεν μένεις και εσύ ικανοποιημένος. Ε, δεν συμβαίνουν μόνο κακά πράγματα στον κόσμο και η λέξη βιωσιμότητα γνωρίζουμε από πού προέρχεται το 1713 ο Κάλοβιτς εξέφρασε για πρώτη φορά αυτήν την αρχή και είναι πολύ απλή η αρχή αυτή διαπίστωσε ότι δεν επιτρέπεται να παίρνουμε περισσότερα από τη φύση από όσα ξαναφυτρώνουν. Και αγαπητέ Μάρτιν Χόισλινγκ, όταν χρησιμοποιούμε το ξύλο, τότε συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Στο Ρέγκενσπουργκ Ε, υπάρχουν ε, πολλά ξύλινα πατώματα τα οποία κανείς ε, δεν, κανένα έντομο δεν έχει φάει μέχρι τώρα. Εδώ και 500 χρόνια υπάρχουν στο Δημαρχείο και στην, Γερμαν... στην Φιλανδία όλο ξύλινα σπίτια είναι. Έτσι λοιπόν μπορούμε να συμβάλλουμε στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, διότι δεσμεύεται το διοξίδιο του άνθρακα. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε όσον αφορά την αναδάσωση. Έχουμε συγχρηματοδοτήσει πρόγραμμα αναδάσωσης στην Βραζιλία και χαίρομαι που υπάρχουν εκεί ωραία νέα δάση. Ε, όταν στηρίζουμε τέτοια προγράμματα θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, φυτεύεται ξυλία που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, διότι αν απλά ε, έχουμε δάση που απλά σαπίζουν, ε, τότε απελευθερώνεται πάλι διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ε, το, την ξυλία που φυτρώνει και υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να βελτιωθεί η εκμετάλλευση της ξυλίας. Θα ήθελα να συμφωνήσω επίσης με τη συνάδελφο Μαριάννα Πιτήρ. Θα πρέπει κατά τους υπολογισμούς να λάβουμε υπόψη μας και την κατάσταση του παρελθόντος. Ε, συμφωνώ με την Ελίσσα Πετκέρστιγκερ ότι η γεωργία και η δασοκομεία δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος, αποτελούν μέρος της λύσης. Ε, και ε, νομίζω μπορούμε να συμβάλλουμε έτσι στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είμαι γενικά αρκετά σκεπτικό όσον αφορά το σύνολο τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή πραγματικά είναι ονειρεμένη μέρα. Συμπίπτουν οι συνεδριάσεις τριών επιτροπών, δύο ψηφοφορίες. Εν πάση περιπτώσει έκανα ό,τι μπορούσα για να έρθω και να πάρω το λόγο γιατί το θέμα της υγιής, αλλαγής χρήσης και δασοκομείας είναι πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη αλλά κυρίως για την πατρίδα μου τη Φιλανδία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, κυρίες Μίλλερ και Κάστιγκερ γιατί πραγματικά στάθηκαν στα πιο σημαντικά τμήματα της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να προβλέπει συμμόρφωση με τους κανόνες. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δάση ως ε, δεσμευτικά του διοξιδίου του άνθρακα και να μην υποτιμούμε το ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό το άρθρο 8 της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί λαμβάνεται ως περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό η περίοδος 1990 μέχρι 2009. Κατά τη γνώμη μου είναι εσφαλμένος ο τρόπος υπολογισμού. Πώς είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Έχουμε δύο διαφορετικά σημεία που θα πρέπει να συμπεριλάβουμε. Στον τρόπο υπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν προβλήματα γιατί δεν εθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν η φόρο διαχείριση των δασών. Υπάρχει μεγάλη αντίφαση στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το ζητούμενο και την ενθάρρυνση και γίνεται πολλής λόγος για τη βιομάζα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Κέστιγκερ που ζητά ο υπολογισμός να εδράζεται σε τωρινά στοιχεία για να καλυφθούν οι αδυναμίες της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα καταθέσω και κάποιες τεχνικές ε, τροπολογίες, πάντως ε, ε, γενικά συμφωνώ με την εισηγητρία και την γνωμοδότηση και πιστεύω ότι η πολιτική ε, για τα δάση θα πρέπει να εξαρτάται από τα κράτη-μέλη και σε αυτά επαφίεται η διακριτική ευχαίρεια της λήψης αποφάσεων. Και θα πρέπει ο κανονισμός ΛΟΥΛΟΥΣΕΦ να ενθαρρύνει μια υφόρο διαχείριση των δασών για να αναπτυχθούν περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαδραματίσουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο ως ε, ε, μέρη του διοξιδίου του άνθρακα. Η πρόταση Λουλουσεφ θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τον ιδιάζοντα χαρακτήρα των ιδιοκτητών και διαχειριστών των δασικών εκτάσεων. Όπως σας είπα θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες για άλλα θέματα, κυρίως ε, για τα προϊόντα της ξυλίας. Θα πρέπει και αυτά να συνυπολογίζονται σε μια ειδική κατηγορία όμως. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Κέστιγκερ φυσικά, λέει ο κύριος Δενανό. Είναι πολύ πλήρης και με πολλά πλεονεκτήματα αυτή η έκθεση. Είναι σαφές ότι ο ρόλος των γεών και της χρήσης τους ε, αποτελεί βασικό στοιχείο στην καταπολέμηση της υπερθερμαστού πλανήτη. Εμείς πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και να έχουμε κοινού κανόνες ακόμα και αν τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο ισχυρίζονται ορισμένοι. Πράγματι τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης αλλά το ίδιο ισχύει και για τις γεωργικές ε, γεές και τα ε, μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι Πρέπει να δοθούν κλιματικές λύσεις και να έχουμε ένα παγκόσμιο όραμα. Η ισορροπία μεταξύ γεωργικών γεών και δασών πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Δεν πρέπει να τα θεωρούμε αντίθετα, αλλά συμπληρωματικά στοιχεία. Αυτό θα πρέπει να καταλήξει σε συστάσεις, επειδή τα κράτη-μέλη πρέπει να διατηρήσουν κάποια κυριαρχία. Όπως είπε ο Νικολά Καπούτο, θα πρέπει να διαφερθούμε και στα, στα προϊόντα από τα δάση. Ε, είναι σημαντικό διότι τα είδη ξύλου διαφέρουν από χώρα σε χώρα ε, και η χρήση διαφέρει. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε λοιπόν τα δάση στην Κροατία, στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στη Γαλλία. Ούτε μπορούμε να συγκρίνουμε την Τάιγκα με τα δάση του Αμαζονίου. Κάθε κράτος λοιπόν πρέπει να μπορεί να έχει τη δική του ερμηνεία με μια βασική κοινή ερμηνεία. Αυτή είναι η ουσία της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Ε, μια και είστε ο εισηγητής τη κατ' ουσία Επιτροπή ΕΜΒΗ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, συντάκτρια την Ελίζα Πέτ Νομίζω ότι έχει συμπεριλάβει σωστά και σημαντικά πράγματα στη γνωμοδότησή της. Θα προσπαθήσω στην ΕΝΒΗ, την επί της αρμόδια επιτροπή, να συμπεριλάβω στην έκθεσή μου πολλά από αυτά που πρότεινε. Αλλά με. Πρέπει να το πω αυτό ανοιχτά. Ε, βλέπω δύο ομάδες σοσιαλιστών εδώ. Άκουσα αυτά που είπε χθε ο συνάδελφος Πρέναν. Όλα όσα πρότεινα εγώ για την δασοκομεία, για την ισχυρότερη συμμετοχή των κρατών μελών, για την ε, τροποποίηση των επιπέδων αναφοράς, ε, αναφέρθηκε ως παράδειγμα η Κροατία, οι συνάδελφοι Αντρίο και Καπούτο θα ήθελα να παρακαλέσω τους δύο αυτούς συναδέλφους την ε, συζήτηση αυτή να την έχουν ε, εντός ε, της ομάδας των ε, σοσιαλιστών. Δεν μπορείτε εδώ να λέτε κάτι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να λέτε το αντίθετο. Προσβλέπω στη συζήτηση εντός της ομάδας των σοσιαλιστών και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω στην έκθεσή μου πολλά από αυτά που ακούστηκαν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δάντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω και να επενέσω το έργο της κυρίας Κέστιγκερ όπως έκανα χθε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το έργο του Νόρμπερτ Λίνς. Επίσης, συμφωνώ με την τήρηση της αρχής επικουρικότητας ό,τι αφορά την πολιτική για τα δάση. Σε ό,τι αφορά το εθνικό επίπεδο αναφοράς, άρθρο 8, συμφωνώ απόλυτα με την διαπίστωση που κάνει η συγγήτρια κυρία Κιώστιγκερ, ε, ε, γιατί ένα επίπεδο που στηρίζεται σε ιστορικά ε, δεδομένα έχει ελλείψεις. Καταρχήν μια ιστορική βάση ε, ουσιαστικά φέρνει σε δυσμενή ε, μεταχείριση τα κράτη που έχουν πρόσφατα τη μια αηφόρη πολιτική και αποθαρρύνει άλλα κράτη από την εφαρμογή τέτοια υφόρου πολιτικής. Επίση, η αύξηση τη εκμετάλλευση των δασών θα υπολογιστεί αρνητικά ταυτόχρονα έχουμε άλλες πολιτικές που εθαρρύνουν και τη χρήση της βιομάζας και την ε, βιώσιμη δέσμευση του άνθρακα. Η ξυλία και τα δάση πληρούν δύο προϋποθέσεις. Θα μπορούσαν ταυτόχρονα να αποτελούν τμήμα της ενεργειακής μας πολιτικής, του ενεργειακού μείγματος όπως λέμε, γιατί το ξύλο ε, είναι μια ανανεώσιμη πηγή ουσιαστικά και επίση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον οικοδομικό κλάδο, στο κατασκευαστικό τομέα, ως ε, πολύ κατάλληλο υλικό που επιτρέπει ταυτόχρονα την ε, βιώσιμη αποθήκευση του άνθρακα. Οπότε δεν, δεν μπορούμε σε μία πολιτική να, να ισχυριζόμαστε κάτι και μετά να το α, ε, καταρρύπτουμε σε άλλη πολιτική. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Είμαστε υπέρ της κυκλικής πολιτικής, της κυκλικής οικονομίας και γι' αυτό συμφωνώ ε, με τον προσδιορισμό εθνικών επιβέδων αναφορά με βάση την τωρινή πολιτική αηφόρου διαχείριση και όχι με βάση ιστορικά δεδομένα που δεν προσαρμόζονται στη σημερινή κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Αλμπερτέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο σύντομες παρατηρήσει. Καταρχάς ο Νόρμπερτ Λίνς είπε ότι ακούει τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και έχει την εντύπωση ότι έχει δύο πολιτικές ομάδες μπροστά του. Άλλωστε είναι σοσιαλιστές και δημοκράτες. Πρόκειται λοιπόν για δύο ομάδες. Και μία ακόμα παρατήρηση. Σας παρακαλώ επαναλάβετε το, του λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητοί, αγαπητές συνάδελφε Ταραμπέλα, ε, αναρωτιέμαι, οι σοσιαλιστές δεν είναι δημοκράτες, αφού τονίζετε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Και δεύτερη παρατήρηση που ξέχασα πριν. Κατά τους υπολογισμούς αυτούς ε, θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη ότι κάποιες ε, χώρες έχουν αναδασώσει σημαντικές εκτάσεις τα τελευταία χρόνια. Ε, στη Γερμανία έχουμε ένα εκατομμύριο περισσότερα εκτάρια δασών από ότι πριν 15 χρόνια. Θα πρέπει και αυτό να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό. Ο κύριος Άγνιου. Σας ευχαριστώ που με επιτρέπετε να δευτερολογήσω. Ο ευρωβουλευτής που πήρε το λόγο πριν τον κύριο ε, μίλησε για ξύλινα σπίτια. Τα δικά σας όμως ε, δεν νομίζω ότι εισέρχονται στο έδαφος. Ε, αυτή είναι η χίλιος πτέρνα όλων των ξύλινων σπιτιών. Τα περισσότερα ξύλινα σπίτια που έχω δει είναι χτισμένα πάνω σε μια βάση, πάνω σε θεμέλια πέτρινα διότι οποιοδήποτε ξύλο θα ε, διασπαστεί μέσα σε 10-15 χρόνια. Καταλαβαίνω ότι στην ε, Σκανδιναβία ε, είναι τόσο δημοφιλή τα ξύλινα σπίτια, αλλά εκεί είναι παγωμένο το έδαφος επί μήνες και αυτό αποτρέπει τα έντομα. Θα πρέπει όμως να εντοπίσουμε ότι το ξύλο είναι οργανικό προϊόν, έχει περιορισμένη ζωή. Είτε λοιπόν θα έχει κανείς το ξύλο που θα φυτρώνει επί 200 χρόνια και κατόπιν θα σαπίσει και θα οδηγήσει σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ή θα γίνει κάποιο ξύλινο προϊόν που επίσης θα σαπίσει εκτός εάν ε, το επεξεργαστούμε με ε, σημαντικά συντηρητικά. Αλλά ποια είναι η ε, δική τους συμβολή στο διοξίδιο του άνθρακα και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στον υπολογισμό. Κάποια στιγμή το ξύλο εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον κύριο Χάιμ από τη Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που ακούω ότι η Επιτροπή Άγκρη συζητά την πρόταση αυτή και ευχαριστώ την εισηγήτρια για τις προσπαθίες της. Να υπενθυμίσω ότι το ζήτημα αυτό συζητείται στο Κοινοβούλιο με τους συνομοθέτες για δεύτερη φορά. Τα κράτη-μέλη ήδη υλοποιούν παρόμοιους κανόνες με αυτούς του κανονισμού αυτού στο πλαίσιο της σημερινής περίοδου δεύτερης, της δεύτερης περίοδου Είναι σημαντικό να πούμε ότι τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό για τους ε, αγρότες ή τους δασοκόμους. Τα κράτη-μέλη υλοποιούν πράγματα τα οποία σημειώνουν καταπληκτική πρόοδο και που συνάδουν με την αηφόρο διαχείριση των δασών και που συμμορφώνονται με την ευημερία του γεωργικού τομέα χωρίς να περιορίζεται η διατροφική ασφάλεια. Οι κανόνες που προβλέπουμε τώρα για την ε, περίοδο 2021 μέχρι 2030 είναι παρεμφερείς με τους σημερινούς. Με την τρέχουσα υλοποίηση τα κράτη-μέλη αποκτούν εμπειρία με τη βελτίωση της παρακολούθησης και του υπολογισμού διαφόρων δραστηριοτήτων στους τομείς αυτούς και για τη γεωργική γη και για την ε, αναδάσωση. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να συμπεριληφθούν οι δραστηριότητες αυτές ε, στο μηχανισμό ευελιξίας ε, από το LULUCF στο στόχο επιμερισμού προσπαθειών. Συμπεριλαμβάνοντας το LULUCF συμπεριλαμβάνουμε 20-30 κλιματικούς στόχους. Είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται ότι οι δύο πλευρέ του ίδιου νομίσματο είναι υπαρκτέ. Από τη μια μεριά έχουμε τι εκπομπέ από τη Γεωργία, αλλά μέσω τη χρήση γη και την καλύτερη δέσμευση άνθρακα στο γεωργικό έδαφο και την αναδάσωση, η Γεωργία μπορεί να αποτελεί κομμάτι τη λύση τελικά. Αυτό να γνωρίζετε ρητά ε, μέσα σε αυτή την ευελιξία που παρέχουμε. Η έκταση της ευελιξίας αυτής ε, κατά κάποιο τρόπο καθορίζεται έτσι ώστε ο γεωργικός τομέας σε τελική ανάλυση να χρησιμοποιεί ε, αποτελεσματικές επιλογές μετριασμού ως προς το κόστος χωρίς να αυξάνεται το κόστος για τον γεωργικό τομέα. Αυτό είναι κατά την άποψή μας πολύ σημαντικό. Ένα άλλο θέμα προς είναι η λογιστική των δασών ε, σε αυτόν τον τομέα, στην πρόταση της Κομισιόν. Να σεβόμαστε απόλυτα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για τις δασικές πολιτικές. Τα κράτη-μέλη βρίσκονται στη θέση του οδηγού. Αυτά υπολογίζουν ε, τις τιμές αναφοράς για τα δάση. Ουσιαστικά την προσέγγιση αυτή την πρότεινα τα κράτη-μέλη στις συζητήσεις, ε, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Τόκιο. Γιατί διότι έτσι τα κράτη-μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικών τους δασών, ε, τη δική τους δομή Ε, κάτι απαραίτητο διότι το πρωτόκολλο του Κιώτο κάποια στιγμή θα διακοπεί και η διακυβέρνηση ε, και η αναθεώρηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτείνει η Κομισιόν ε, θα βοηθήσει να προσδιοριστούν ε, αυτές οι τιμές. Το τι θα γίνει ακριβώς θα συζητηθεί πιο λεπτομερώς. Επιπροσθέτως η πρόταση αναγνωρίζει σαφώς τα πλεονεκτήματα της χρήσης των δασικών προϊόντων, ε, της ε, διαχείρισης ε, των διαφόρων γεών από τη Γεωργία και πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι η πρόταση της Κομισιόν συνάδει απόλυτα με τις αρχές αηφόρου διαχείρισης των δασών δίνει τη δυνατότητα για ευημερία της βιολογικής οικονομίας και συμμορφώνεται απόλυτα με τη διατροφική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Okay. Μάλιστα. Η μας τώρα, κυρία Κέστιγκερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πολλές ε, θετικές παρατηρήσεις και θα ήθελα να συμφωνήσω με όλα όσα υπόθηκαν κατά της επιπλέον γραφειοκρατίας, διότι το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό. Έχουμε εκατομμύρια ιδιώτες, ε, ιδιοκτήτες ε, δασικών εκτάσεων ε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να τους λάβουμε υπόψη μας και όχι να αρχίσουμε να ρυθμίζουμε πράγματα τα οποία τελικά δεν θα λειτουργήσουν. Ε, μία σύντομη παρατήρηση προς τον κύριο Φλάναγκαν. Ε, συμφωνώ όσον αφορά τους ε, υγροβιότοπους και ε, τους τυρφώνες. Ε, άλλωστε, δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε κάποια συγκεκριμένα γεωργικά μοντέλα. Αντιθέτως, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι έχει γίνει στον τομέα της γεωργίας, σε ποια περιβαλλοντικά προγράμματα λειτουργούν καλά και θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Όσον αφορά τους υγροβιότοπους, αυτό που ανέφερε ο κύριος ε, Φλαναγκάν, ε, δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην πρόταση Λουλουσιεφ. Έχουν εξαιρεθεί και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχω επίσης ε, πολύ καλά νέα για τον κύριο Άγνιου. Ε, τα ξύλινα σπίτια ε, δεν είναι πια όπως ήταν. Τον προσκαλώ στην Αυστρία όπου ε, έχουμε το 2018 θα ολοκληρωθεί υβριδικό κτίριο 48 ε, ορόφων ε, και η σύγχρονη τεχνολογία ξύλου αντικαθιστά παλαιά ορυκτά υλικά. Και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ληφθούν ε, πολύ περισσότερο υπόψη όλες αυτές οι πτυχές ε, και αυτή άλλωστε είναι η κατεύθυνση του μέλλοντος. Στην Μαριάννα Πέτυρ. Να πω ότι έχω διαγράψει το χρονικό διάστημα μέχρι το 2009, διότι για τους λόγους που υπόθηκαν ε, πιστεύω ότι είναι σωστό να μην επιτρέψουμε να υπάρχει οποιαδήποτε αδικία εδώ. Όσον αφορά τη στρατηγική για την ε, βιοοικονομία και την ε, βιοπικιλότητα, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ, να ληφθούν υπόψη. Θα αφήσουμε λοιπόν ε, τις ιστορικές περιόδους λίγο πολύ ως έχουν. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Χόισλινγκ, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Η εμπορία εκπομπών ρυθμίζεται στο σχετικό σύστημα και Υπάρχει εδώ ένα μικρό λαθάκι. Τα δάση είναι ε, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ε, αποτελεί αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό η δασοκομεία και η δασοπονία να συνεχίσουν να αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η ε, εκπρόσωποι της Κομισιόν επίσης ε, έχουν πει σαφώς εδώ τη γνώμη τους. Δεν θα λειτουργήσει το σύστημα αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε ε, ευρωπαϊκό. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ουσιαστικό θέμα η αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι δασοκόμοι γνωρίζουν ακριβώς τι θα πρέπει να κάνουν ώστε και οι επόμενες γενιές να μπορούν να υποφεληθούν ε, από αυτήν την ε, πηγή. Και εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε στεναρά αυτήν την ιδέα του one size fits all. Σημαντικό πάντως είναι ότι μεγαλώνουν περισσότερα νέα δάση από αυτά που αποψηλώνονται και Η Επιτροπή Γεωργίας ε, πιστεύω ότι θα αποτελέσει δυνατή φωνή υπέρ των δασών και υπέρ των δασοκόμων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Φαντάζομαι θα μας προσκαλέσετε όλους ε, στην Αυστρία και τον κύριο Άγνου ιδιαιτέρως για να δει αυτό το καταπληκτικό νέο κτίριο. Η προθεσμία για τις τροπολογίες λήγει στη 1 η ώρα 27 Μαρτίου. Ε, και θα ήθελα να μας στείλετε και γραπτό σε ένα σημείωμα με τα, αυτά τα χρήσιμα επιχειρήματα. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να μας το στείλετε γιατί θα τα αξιοποιήσουμε και στις περαιτέρω μας συναντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, οπότε δεν χρειάστηκε να σας περιορίσω. Ολοκληρώνουμε την δημόσια συνεδρίασή μας. Μετά από μια σύντομη τεχνική διακοπή θα αρχίσουμε εντός ολίγου, μετά από τρία λεπτά μια τεχνική, ένα τεχνικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα περάσουμε συνεδρία των συντονιστών.